Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατανοώ ότι η ώρα περνάει και πρέπει να τελειώσετε. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις σας, γιατί νομίζω ότι επιβεβαίωσαν την πραγματογνωμοσύνη σας. Ε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και στην Επιτροπή Βιομηχανίας και Έρευνας. Επομένως, διαπιστώσαμε για μία ακόμα φορά τις γνώσεις σας αλλά και την αφοσίωση που έχετε όσον αφορά ε, τα ζητήματα αυτά που μας ε, απασχολούν. Ξέρω ότι εργάζεστε ε, πολλά χρόνια εδώ και πολλά χρόνια ε, για τα θέματα αυτά και ε, έχετε πραγματικά επιτύχει πάρα πολλά. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή η επιτυχία και η σε αντιμετώπιση των ζητημάτων συνεχιστεί και τα επόμενα πέντε χρόνια στη νέα θητεία του Κοινοβουλίου. Προσπάθησα να σας εξηγήσω ποια είναι τα κριτήρια ε, ε, με τα οποία κρίνουν και εμάς και την Επιτροπή δηλαδή και τους, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι πολίτες και επ' αυτόν να βασίσω και τους πυλώνες εργασίας μου Θέλουν οι πολίτες λοιπόν καθαρή ε, προσιτή ενέργεια. Αυτό πρέπει να τους δώσουμε. Επίσης ζητούν αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη και ε, ασφάλεια όσον αφορά την ε, ενέργεια. Όσον αφορά τώρα την ανάπτυξη θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να δημιουργήσουμε νέες θέσει εργασία. Αντιμετωπίζει η Ευρώπη πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, σκληρό άγριο ανταγωνισμό σε αυτόν τον νέο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Θα πρέπει να το κάνουμε ε, με τρόπο σωστό, ε, έτσι όπως εμείς καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη, δηλαδή με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον ε, και με διατήρηση των κοινωνικών προτύπων. Φυσικά δεν υπάρχουν εύκολες ερωτήσεις σε αυτά τα δύσκολα ερωτήματα και ε, νομίζω ότι ο τρόπος που θα μας αντιμετωπίσουν οι πολίτες, ε, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι κριτές, ε, θα είναι και ο, τρόπο, θα είναι και ο οδηγός μας σε αυτήν την, την πορεία. Πιστεύω πάντως ότι η Ευρώπη είναι στη σωστή θέση, έχει όλα αυτά τα απαραίτητα συστατικά έτσι ώστε να προχωρήσει και πιστεύω ότι εάν καταβάλουμε προσπάθειες από κοινού θα καταφέρουμε να καλύψουμε τις διαφορές. Ξέρετε ότι στην παρούσα θητεία της Κομισιόν ήμουν υπεύθυνος και για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο ε, και δούλεψα πάρα πολύ, συνεργάστηκα πολύ με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, την Νομική Επιτροπή, πολύ στενά συνεργάστηκα με τον ε, Πρόεδρο Μπουζέκ στη διάσκεψη των ε, Προέδρων. και την εποχή βεβαίως που ήταν και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως εγώ είμαι θερμός υποστηρικτής της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων, είμαι θερμός υποστηρικτής του δομημένου διαλόγου αλλά και της ε, σωστής ε, αξιολόγησης, προετοιμασίας ε, της εργασίας και όσον αφορά και εάν εγκρίνεται την νέα μου θέση θα συνεχίσω την συνεργασία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο θα είμαι πάντα έτοιμος να έρθω εδώ οποτεδήποτε μου το ζητήσετε να συζητήσω μαζί σας, να ανταλλάξουμε απόψεις ε, και βεβαίως και σε επίσημο αλλά και σε προσωπικό επίπεδο με τον καθένα από εσά θα ήθελα να έχω ε, την ε, επαφή αυτή η οποία θα μας συντροφέψει για τα επόμενα πέντε χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και εάν ε, τύχω τη στήριξή σας ε, δεσμεύομαι να συνεχίσω την καλή συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Uh, σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, κύριε Υποψήφια Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε και για τις δηλώσεις σας ε, και για τις απαντήσεις και για αυτές τις πέντε μέρες σκληρής δουλειάς που κάνατε έτσι ώστε να προετοιμαστείτε για την ακρόαση αυτή όλοι οι συνάδελφοι που είναι εδώ σας ευχαριστούν. Σας ευχαριστώ και εγώ αγαπητοί συνάδελφοι γιατί έχετε υπομονή αλλά έχετε και πάθος. Είσαστε παθιασμένοι με τα θέματα. Και σε ό,τι αφορά την Ήτρε, οι συντονιστές για την συνάντηση αξιολόγησης θα συναντηθούν αύριο στις 9.30. Με, μετά θα γίνει κίνημα στις συνεδρίαση με την Επιτροπή Ήτρε ε, Ευχαριστώ πολύ και τον Τζάνι Λαβία. Και εγώ ευχαριστώ. Αύριο θα έχουμε τη συνάντησή μας στις 9 και μετά θα συναντήσουμε και τους συντονιστές της Επιτροπής Ήτρε για την τελική μας αξιολόγηση. Ε, καλή όρεξη, λίγο αργά είναι, αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε. Γεια σας.